Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω να καθίσετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη ε, τιμή για μένα να μπορούμε να καλωσορίσουμε εδώ σήμερα τον ε, πρόεδρο της Πορτογαλίας, τον κύριο Καβάκο Σίλβα. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια περίεργη έκτακτη κατάσταση με την εξής έννοια. Έχουμε δύο προσωπικότητες ε, που ε, συμμετείχαν ουσιαστικά στο να εισέλθει η Πορτογαλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άσκησαν ε, τεράστια επιρροή και σήμερα οι άνθρωποι αυτοί έχουν διαφορετικές ε, θέσεις από ό,τι είχαν τότε. Ο κύριος ε, Καμπάκο Σίλβα τότε ήταν ε, ο Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας και ο κύριος Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο τότε ήταν υφυπουργό, αργότερα υπουργό εξωτερικών και αργότερα και πρωθυπουργό της Πορτογαλίας αλλά οι δύο αυτοί άνθρωποι σε μια σημαντική φάση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ε, κατήχαν ε, καθοριστικά αξιώματα στη χώρα του. Φαντάζομαι λοιπόν ότι χαίρονται και οι δύο που βρίσκονται σήμερα εδώ με διαφορετικά αξιώματα και ξανά συναντιόνται. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν θερμά κύριε Καβάκο Σίλβα, σας καλωσορίζουμε θερμά κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής ε, και καλωσορίζω θερμά και όλους τους συνεργάτες του κύριου Καβάκο Σίλβα. Κύριε Καβάκο Σίλβα, κύριε Πρόεδρε σας δίνω το λόγο. Κύριε... Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση να απευθυνθώ στο σώμα σας με τιμά. Σέβομαι βαθιά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον ρόλο του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερα σε προηγούμενη παρουσία μου εδώ το Σεπτέμβριο του 2007, γνωρίζω καλά τις δράσεις και τη συνεισφορά του Κοινοβουλίου στην διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δεν ξεχνώ την ειλικρινή υποστήριξη που έλαβα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Πρωθυπουργός κατά, τις, κατά τη διάρκεια της περίοδου που ηγήθηκα της ε, πρώτης Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου το 1992. Με ικανοποίησή μου υπογραμμίζω την μεγάλη εξέλιξη του Κοινοβουλίου από την εποχή του Μάστριχτ και μετά. Η συνθήκη της Λισαβόνας εδραίωσε πολύ σωστά την, το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου ως συνομοθέτη μαζί με το Συμβούλιο. Πρόκειται για μια επιλογή που καθιστά τη λήψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο δημοκρατική και εμβαθύνει ε, την ε, πολιτική κουλτούρα στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν το καλύτερο σημείο εδώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις για πράγματα τα οποία θεωρώ επίγοντα και επίκαιρα για τους ε, πολίτες μας και τα κράτη μας σε αυτή τη φάση του ευρωπαϊκού σχεδίου του ευρωπαϊκού οράματος. Τις τελευταίες ε, δεκαετίες η ευρωπαϊκή ιδέα ε, ε, χτίστηκε πάνω σε, μια πολιτική, σε ένα πολιτικό οικοδόμημα μοναδικό και μοντέλο για πολλούς. καταρρίχθηκαν τα σύνορα, δημιουργήθηκε η ελευθερία της κυκλοφορίας των, των ατόμων, υποστηρίχθηκε ο πολιτισμός, η γνώση, η νέα αγορά, δημιουργήθηκε η νέα αγορά. Είμαστε το μεγαλύτερο οικονομικό μπλοκ στον κόσμο και βέβαια έχουμε και το ενιαίο νόμισμα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι η έμπνευση ε, και οι επιτυχίες μας ε, δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν ως δεδομένα. Η οικονομική ανάπτυξη είναι πολύ συχνή και πολλές χώρες βρίσκονται σε ύφεση. Η ανεργία είναι ψηλή και μια, πραγματικά δραματική, μια δραματική πραγματικότητα. Ε, έχουμε σημαντικές προκλήσεις και χρειαζόμαστε αποτελεσματικές απαντήσεις. Δεν μας εκπλήσει λοιπόν που ε, χάνουμε σε μεγάλο βαθμό, μάλλον ε, υπάρχει ε, μεγάλο ρήγμα μεταξύ των αποφάσεων, μεταξύ αυτών που παίρνουν τι αποφάσεις και των πολιτών. Πριν από 28 χρόνια, στις 12 Ιανουαρίου του 1985, η Πορτογαλία υπέγραψε ε, στο μοναστήρι των Ζερόνιμους στην ε, Λισαβόνα τη δέσμευσή της να ενταχθεί στην, ε, στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Η ένταξη της Πορτογαλίας αποτέλεσε το, την κορύφωση του εκδημοκρατισμού της χώρας και συνσέφερε αποφασιστικά για την ανάπτυξη της χώρας. Από τότε η Πορτογαλία συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η Πορτογαλία έφερε στην Ευρώπη την ιστορική τη σκληρονομιά, ε, το, τη σφραγίδα του Ατλαντικού Διαλόγου, τη μαγκοσμιότητα της γλώσσας και της κουλτούρας της. Ε, έχουμε στενούς δεσμούς με την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Ε, και ομογένεια σε όλα τα μέρη του κόσμου. Φέραμε επίσης την ε, εδραίωση της, ε, του διεθνούς χαρακτήρα της ε, κοινότητας των χωρών που μιλούν την πορτογαλική γλώσσα και όλοι αυτοί είναι παράγοντες που συνεισφέρουν στο συνολικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, όπως γνωρίζετε, οι Πορτογάλοι ζουν μια ε, έντονη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση με όλες τις βαριές συνέπειες, κοινωνικές συνέπειες που φέρνουν αυτές οι κρίσεις. Τα τελευταία χρόνια ε, ήταν για τη χώρα μου από τα πιο περίπλοκα που έχουμε ζήσει τα, στην, στην πρόσφατη ιστορία μας. Από το μέσο του 2011 ε, κάνουμε μια σημαντική προσπάθεια οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ε, προσαρμογής ε, στο πλαίσιο του ε, προγράμματος το οποίο συμφωνήσαμε με τα διεθνή θεσμικά όργανα. Η διαδικασία εξ, δημοσιονομικής εξυγίανσης προχωράει. Παρόλο ότι το πλαίσιο στο οποίο κινούμε είναι πολύ πιο αρνητικό από αυτό που είχε προβλεφθεί αρχικά και παρόλο το ασύμετρο σοκ το οποίο ζούμε. Στη χώρα μου ε, η ύφεση έχει οδηγήσει, ε, διαρκεί εδώ και 10 τρίμηνα. Η ανεργία έχει φτάσει στο 17,7% και η ανεργία των νέων στο 42%. Ε, αυξάνεται επίσης σε επικίνδυνο βαθμό η φτώχεια. Απαιτούνται σημαντικές θυσίες από τους Πορτογάλους πολίτες, οι οποίοι έχουν δείξει αίσθημα ευθύνης έχουν ενισχύσει τους δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ τους και αλληλοβοηθούνται με τρόπο που να μετριάζονται οι πιο δραματικές καταστάσεις. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, αυτή η κρίση κατέστησε πιο σαφή το βαθμό αλληλοεξάρτησης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα και της ε, Ευρωζώνης ειδικότερα. Είναι το λογικό αποτέλεσμα Τη ολοκλήρωση την οποία έχουμε πετύχει. Δεν είναι δυνατόν να διαχωρίσουμε την κατάσταση σε ένα κράτος μέλος από αυτήν στο, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Με δύο λόγια είμαστε μια ένωση και όχι ένα συσσωμάτωμα κρατών ή αγορών. Και αυτό δημιουργεί μεγάλη διαφορά όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε την πραγματική σημερινή κατάσταση και να αποφασίσουμε ποια είναι η κατάλληλη απάντηση. Τα τελευταία δύο χρόνια πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε σημαντικές προσπάθειες σε ό,τι αφορά της, ε, την υποστήριξη των αναγκών χρηματοδότησης των κρατών μελών που ε, ε, έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και επίσης την εφαρμογή κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας και επιτήρησης και στην εμβάθυνση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Η Ευρωπαϊκή Αντική Τράπεζα ανακοίνωσε την ε, δυνατότητα να παρεμβαίνει χωρίς όριο στη δευτερογενή αγορά κρατικού χρέους. Ε, πρόκειται για ένα σημαντικό πλαίσιο το οποίο απέκρουσε τις ε, κερδοσκοπικές προσπάθειες στη ζώνη ευρώ. Παρόλε τι θετικέ αυτέ εξελίξει, πρέπει να αντιληφθούμε και να παραδεχτούμε ότι η κρίση κατέδειξε τι της τη Ένωση πέραν της αργής και υπερβολικά ήπιας απάντησης στην κρίση του ευρώ, ε, η μεγαλύτερη αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βρισκόταν και βρίσκεται στην ε, πρόθεση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Το 2012 η Ευρωζώνη είδε το ΑΕΠ τη να συρρυκνώνεται κατά 0,6% και οι προβλέψεις για το μέλλον είναι ότι θα έχουμε αρνητική ανάπτυξη και το 2013. Η ανεργία στην ε, Ένωση αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία πέντε χρόνια. 26 εκατομμύρια είναι πλέον οι άνεργοι, εκ των οποίων 5 εκατομμύρια 700.000 είναι νέοι. Η Ευρωζώνη βρίσκεται στο έκτο ε, συνεχές τρίμηνο ε, ε μείωσης του ΑΕΠ και το 8ο τρίμηνο μείωσης των επενδύσεων η τάση είναι αντίθετη στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιαπωνία. Εδώ και υπερβολικά πολύ χρόνο ε, εστιαστήκαμε στην λιτότητα για να διορθωθούν οι ανισορροπίες ε, ε, στα, δημόσια οικονομικά, βάζοντας σε δεύτερο πλάνο την οικονομική ανάπτυξη. αργήσαμε στις ε, μεταρρυθμίσεις και σε πολλά κράτη-μέλη οι ε, επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα στη χρηματοδότησή τους. Ε, η εμπιστοσύνη μειώνεται και αυτό ε, υποσκάπτει τις επενδύσεις. Η μείωση της εσωτερικής ζήτησης στο σύνολο της Ευρωζώνης οξύνει τα προβλήματα που για παράδειγμα έχει η Πορτογαλία στο να επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους και αυξάνει την ύφεση και την ανεργία. Όταν στις ε, χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα εξυγίανσης ε, προστίθενται ε, πολιτικές λιτότητας και συσταλτικές πολιτικές σε άλλα κράτη-μέλη, η συνέπεια είναι ύφεση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που βλέπουμε σήμερα. η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική σε άλλα οικονομικά μπλοκ που ακολουθούν επεκτατικές οικονομικές πολιτικές. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι δεν υπήρξε έλλειψη οράματος, ε, ούτε και έλλειψη προειδοποιήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή και από το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά, αφορά το στόχο της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ε, ε, που θα πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι με την διόρθωση των δημοσιονομικών. Για παράδειγμα, το Δεκέμβριο του 2011 ο πρόεδρος τη Επιτροπή. Ε, απευθυνόμενο σε αυτό εδώ ακριβώ το Κοινοβούλιο είπε δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε, να οικοδομήσουμε μια ε, οικονομική ένωση μόνο πάνω στην πειθαρχία και τις κυρώσεις. Χρειαζόμαστε επίσης και μια Ευρώπη ανάπτυξης και απασχόλησης. Και δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ε, τους αναρρύθμιτες περιπτώσεις οι οποίες από την αρχή της κρίσης εδώ, σε αυτήν εδώ την ε, Ολομέλεια ε, πολλοί βουλευτές από όλες τις ε, πολιτικές οικογένειες συμπεριλαμβάνουν και των Πορτογάλων συμπεριλαμβανομένου και εσάς κύριε Πρόεδρε Σούλτς προειδοποίησατε, προειδοποίησαν για την ανάγκη να μην ξεχάσουμε και αυτή την προτεραιότητα. Η δισταγμή των πολιτικών σε επίπεδο κράτους μέλους όμως καθυστέρησαν την αναγνώριση ότι ο γεγονότος ότι τα οικονομικά, χρηματοοικονομικά προβλήματα κάποιων χωρών επηρεάζουν όλους και ότι η κρίση της Ευρωζώνης δεν λύνεται μόνο με την προώθηση πολιτικών λιτότητας στα κράτη που έχουν υπερβολικά ελλείμματα. Στα, σε ό,τι αφορά τις χώρες που βρίσκονται σε προγράμματα εξυγίανσης θα μπορούσε να έχει αναγνωριστεί πιο νωρίς το πλεονέκτημα ε, των αυτόματων σταθεροποιητών Δηλαδή, να μην επιμείνουμε στην αύξηση των προσπαθειών δημοσιονομικής εξυγίανσης μόνο γιατί ε, η οικονομική χρήση μειώνει τα δημοσιονομικά έσοδα. Οι, οι, οι οικονομίες μας αλλοεξαρτώνται και αυτό απαιτεί από τα κράτη-μέλη να συντονίζουν τις πολιτικές τους. Οι χώρες πια δεν είναι ικανές από μόνες, τις, από μόνες τους, η καθεμία αναλύουν τα προβλήματά τους. Από την άλλη μεριά όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμα δεν έχουμε τα κατάλληλα μέσα για να ε, κάνουμε πραγματικότητα αυτό το αποτελεσματικό συντονισμό. Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση. Τα μέσα που είχαμε στο παρελθόν δεν είναι επαρκή έτσι ώστε η Ευρώπη να απαντήσει, να ανταποκριθεί στα ερωτήματα και στα προβλήματα του σήμερα και να προετοιμάσει το μέλλον. Χρειαζόμαστε να περάσουμε σε μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση με όλες τις πτυχές, τραπεζική, δημοσιονομική, οικονομική. Αυτό θα πρέπει να είναι το βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, είδαμε κάποιες σημαντικές συνεισφορές προς αυτή την κατεύθυνση, για την, δηλαδή για την καινούργια φάση στην οποία πρέπει να μπει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Για παράδειγμα, η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια βαθιά και αυθεντική ε, Ευρωπαϊκή και Οικονομική Ένωση. Επίσης, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεθείτε στο ύψος των περιστάσεων ε, και θα ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Κύριε Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι προβλεφτές. Όπως η επιτυχία της Ευρώπης είναι σημαντική για την Πορτογαλία, έτσι και η επιτυχία της Πορτογαλίας είναι θεμελιώδης σημασία για την επιτυχία της Ευρώπης. Η Πορτογαλία ε, δέχεται, στηρίζεται στην υποστήριξη των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων τη. Ε, ιδιαίτερα στην πρόθεση οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόληση, γιατί αυτέ είναι πολύ σημαντικέ για να επιτύχουμε το στόχο. Χρειάζεται να βελτιώσουμε τι συνθήκε χρηματοδότηση τη οικονομία ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έτσι ώστε είτε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε τα διορθωτικά ταμεία ε, να παίξουν το ρόλο που τους αξίζει, ε, το ρόλο που έχουν. Ε, παράλληλα, είναι σημαντικό το, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, να δώσει μια απάντηση έτσι ώστε να λειτουργήσουν καλύτερα ξανά οι μηχανισμοί διακίνηση του χρήματο σε όλη την Ευρωζώνη. Είναι πολύ σημαντικό να τεθεί σε γρήγορη λειτουργία η, Ευρωπα... Τραπεζική Ένωση για να καταπολεμήσουμε τον κατακαιρματισμό των ε, αγορών, των χρηματαγορών έτσι ώστε η χρηματοδότηση των οικονομιών να γίνεται με ίδιους και ισόρροπους όρους. Είναι απολύτως απαραίτητο να ελαφρύνουμε το υπερβολικό κόστος ε, πιστώσεων, ε, των πιστώσεων που δίδονται στις ε, επιχειρήσεις συγκεκριμένων χωρών όπως η Πορτογαλία το κόστος του χρήματος ε, για πολλές επιχειρήσεις στην Πορτογαλία είναι πολύ ψηλότερο από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κάτι βέβαια που πλήττει την, την ανταγωνιστικότητά τους, επηρεάζει τις αποφάσεις ε, επενδύσεων ε, και προφανώς δημιουργεί αίσθηση αδικίας. Από την άλλη μεριά, είναι σημαντικό οι χώρες που βρίσκονται σε προγράμματα εξυγίανσης να μπορούν να έχουν κίνητρα ε, και ευρωπαϊκή υποστήριξη για τις ε, διαστοτικές αλλαγές που πρέπει να λάβουν χώρα στην, ε, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Για παράδειγμα, να μπορούν προσωρινά να έχουν πρόσβαση σε ένα ειδικό καθεστώς που θα τους επέτρεπε να δίδουν φορολογικά κίνητρα και φοροαπαλλαγές στις επενδύσεις στον τομέα των ε, διαπραγματεύσιμων ε, αγαθών. Δύο λόγια για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κατανοώ, αλλά συμμερίζω πιο πολύ από το ότι κατανοώ, την απογοήτευση ε, πολλών εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο για την έλλειψη φιλοδοξίας από πλευρά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παρ' όλα αυτά, και γι' αυτό μάλλον, γι' αυτό ζητώ να καταλήξουν σύντομα οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Μια άλλη απέτηση της επιτυχίας Πορτογαλίας είναι η πλήρης επιστροφή στις αγορές. Αυτό θα αποτελούσε και ένδειξη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης, συνεπώς θα αύξανε και τις επενδύσεις στη χώρα μου. Τα πρώτα βήματα έγιναν με επιτυχία. Ε, με, ε, με τα ομόλογα, τα πενταετή και δεκαετή ομόλογα ε, που εκδώσαμε φέτος. Αλλά είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να έχουμε την υποστήριξη των ευρωπαϊκών θεσμών. Ε, είναι επίσης πολύ σημαντικό ε, που αυξάνεται το αυξάνονται, διευρύνονται οι προθεσμίες αποπληρωμής των ομολόγων μας. Σα υπενθυμίζω το συμβιβασμό, το, την δέσμευση που είχαν υπογράψει οι αρχή κρατών κυβερνήσεων τη Ευρωζώνη τον Ιούλιο του 2011 σε μια δήλωσή του ε, και την επανέλαβαν τον επόμενο Οκτώβριο. Είπαν, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να, να ε, υποστηρίζουμε τις χώρες που βρίσκονται σε προγράμματα μέχρι ε, να ανακτήσουν αυτές οι χώρες την πρόσβασή τους στην αγορά υπό την προπόθεση ότι ε, εκτελούν επιτυχώς τα προγράμματά τους. Η διευκρίνηση του πώς θα υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση θα συνεισφέρει έτσι ώστε οι χώρες μας να επιστρέψουν στις αγορές. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, η ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα οικοδομήθηκε επί πολλούς αιώνες ε, μοιραζόμαστε κοινούς, κοινές αξίες, κοινά ιδανικά, κάτι που μας ε, ξεχωρίζει ε, ως χώρο δημοκρατίας και ελευθερίας. Η Ευρώπη είναι ένας χώρος στον οποίο θέλουν πολλοί να ζήσουν. Και όχι μόνο για οικονομικούς λόγους. Γιατί εξασφαλίζουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, γιατί είμαστε ένας προορισμός ελευθερίας και δικαιοσύνης. Μετά από, μια, από ένα παγκόσμιο πόλεμο που έπληξε βαθιά την Ήπειρό μας ε, και κόστισε εκατομμύρια ζωές, ε, έγινε δυνατή μια βαθιά ε, ένωση ανάμεσα στα κράτη και τους λαούς μας. Αν δεν υπήρχε αυτή η ένωση, η κίνδυνη καινούργων, καινούριων τραγωδιών ε, δεν θα εξαφανίζονταν από τον οριζοντά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σχέδιο ειρήνης, όπως ε, ανέφερε πριν από λίγο καιρό η Επιτροπή Νόμπελ. Αυτοί που δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρο ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας ε, ε, ξεκίνησαν ένα δρόμο το οποίο εμείς εδώ και πολλές δεκαετίες περπατάμε. Είναι η κοινή αγορά στην Ευρώπη η οποία οδήγησε στην Οικονομική Νομισματική Ένωση. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ο ε, προορισμός, συλλογικός προορισμός των νέων μας που επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθεροι, χωρίς σύνορα. Και οι νέες γενιές στην Ευρώπη δεν θα δεχτούν να ζήσουν με διαφορετικό τρόπο, ούτε να ζήσουν σε διαφορετικό κόσμο. Εξ ονόματος της ειρήνης, αποφασίσαμε να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για μια Ευρώπη ελεύθερη, πιο δυνατή ε, πιο συνεκτικοί και πιο αλληλέγγυοι. Είμαστε Ευρωπαίοι λόγω της ιστορίας μας, αλλά κυρίως είμαστε Ευρωπαίοι γιατί το επιλέξαμε και ζούμε, ε, δημιουργούμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση για την οποία είμαστε περήφανοι. Ε, δεν ήταν εύκολος αυτός ο δρόμος και θα ήταν ε, σημαντική υποχώρηση για την Ευρώπη αν εγκαταλείπαμε αυτό το πνεύμα μιας σταθερής ένωσης με κοινά ιδανικά, με αλληλεγγύη, με θεμελιώδεις αρχές και ε, μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα μας δίνει ισχύ και δύναμη ε, στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Ε, σε αυτή το πλαίσιο η αλληλεγγύη αποτελεί πολιτική, πολιτικά απαραίτητη δράση και όλοι οι Ευρωπαίοι Είμαστε πάνω απ' όλα Ευρωπαίοι και ε, στηρίζουμε το κοινό μας συμφέρον. Αυτή η ευρωπαϊκή κρίση είναι οικονομική και χρηματοοικονομική, αλλά ταυτόχρονα είναι και κρίση δημοκρατική ε, ε, δημοκρατικής νομιμοποίησης. Όλο και περισσότερο οι ευρωπαϊκοί λαοί απομακρύνονται από τους ηγέτες τους και υπάρχουν ανησυχίες ότι το ευρωπαϊκό project δεν κινητοποιεί τους νέους ε, όπως παλιά. Η κρίση δημιούργησε εθνικούς εγωισμούς, ε, τους οποίους θεωρούσαμε ότι είχαμε ξεπεράσει. Αντίθετος με το, με το πνεύμα που ε, χαρακτήριζε την αρχιτεκτονική της Ευρώπης εδώ και δεκαετίες, την οποία εμείς είχαμε φανταστεί ως χώρο ελευθερίας και δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 26 εκατομμύρια ανέργους και η κρίση στην Ευρώπη απαιτεί μια λύση πραγματικά ευρωπαϊκή. Μια λύση ευρωπαϊκή δεν είναι όμως μόνο οικονομική ή χρηματοοικονομική. Χρειάζεται πάνω απ' όλα μια κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική λύση που θα ανταποκρίνεται στις ε, ανησυχίες, θεμητές ανησυχίες των λαών της Ευρώπης είναι ο μόνος τρόπος για να καταπολεμήσουμε, να νικήσουμε μια κρίση εμπιστοσύνης και να ενισχύσουμε την δημοκρατική νομιμοποίηση. Το 2013 έχει κηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. Το 2004 θα λάβουν χώρα εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα αποτελέσουν προφανώς ένα τεστ, μια δοκιμασία για την κινητοποίηση των πολιτών μας. Για να εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη των λαών της Ευρώπης δεν αρκούν ρητορικές δηλώσεις ε, ή δηλώσεις προθέσεων. Αν θέλουμε οι πολίτες να πιστέψουν και να εμπιστευτούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, πρέπει να λαμβάνονται τολμηρές αποφάσεις που θα αποδεικνύουν την αυθεντικότητα αυτού του συλλογικού project. Την αυθεντικότητα των συμφερόντων και των αξιών του της κοινωνικής μεθόδου, με λίγα λόγια. Δεν μπορούμε να χάσουμε περισσότερο χρόνο. Αυτή τη στιγμή, το 2013, θα πρέπει να ικανοποιήσουμε την ελπίδα των 6 εκατομμυρίων νέων που δεν έχουν δουλειά. Το να γιορτάζουμε το Ευρωπαϊκό Χρόνο ε, του πολίτη σημαίνει ότι στοιχηματίζουμε στην οικονομική ανάπτυξη και στην καταπολέμηση ανεργίας. Μόνο έτσι μπορούμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη στο, ε, στο ευρωπαϊκό σχέδιο, στο σχέδιο μιας Ενωμένης Ευρώπης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως αναφέρει η δήλωση Σούμαν, η Ευρώπη δεν θα γίνει διαμιάς Ούτε και όλοι μαζί. Χρειάζονται ε, συγκεκριμένες επιτυχίες, συγκεκριμένα κατορθώματα ε, που βασίζονται σε μια στην, ε, αλληλεγγύη στην πράξη. Ε, είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε. Εξ ε, μια πραγματικής αυθεντικής αλληλεγγύης ήρθε η στιγμή να δείξουμε συγκεκριμένες επιτυχίες στους πολίτες μας, έτσι ώστε η Ευρώπη να παραμείνει χώρος ε, ελπίδας όπως ακριβώς θελήσαμε να τον οικοδομήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε για όλα αυτά που μας είπατε. Κυρίες και κύριοι, φαντάζομαι ομιλώ εκ μέρους όλων ε, ευχαριστώντας τον κύριο Καβάκο